Κόλλιο μπορούμε να την εγκρίνουμε. Δεν βλέπω να έχει κανείς κάποια πρόταση. Ανακοινώσει του Προέδρου. Διαδικαστικά. Καταρχάς, όπως ξέρετε, έχουμε την ε, συνεργασία επί τη βάση του, κανόνου, του κανόνα 55 για τις εκθέσεις ίδιας πρωτοβου... πρωτοβουλίας. 55 Δεν ξέρω, εσείς είστε 56, εμείς είμαστε 54, άρα μέσος όρος 55 για τον κανόνα. Ευχαριστώ, Βίκη. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Βεβαίω είναι πολύ καλή η συνεργασία μας μέχρι στιγμής και κυρίως ε, η κυρία Φόρντ, η κυρία Βίλκουνεν και ο κύριος Ζεβάν ήταν συνεισηγητές, δυστυχώς μετά τις γαλλικές ε, εκλογέ δεν είναι εδώ, γιατί ακόμα έχει διάφορες δυστηριότητε στη Γαλλία. Και να σας πω ότι σήμερα θα δούμε τις τροπολογίες. 462 τροπολογίες υπευλήθησαν για το σχέδιο έκθεσης. η ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της μεικτής Επιτροπής, της μεικτής Συνεδρίας των δύο ε, ε, Επιτροπών, θα γίνει στις 18 Μαΐου στο Στρασβούργο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Online performance και η ψηφιακή ενιαία αγορά προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη. Έχουμε την κυρία Βίρκουνεν και τον κύριο Ζουβάν για να τους ως συζητητές και θα ακούσουμε την κυρία Φόρντ αρχικά να κάνει κάποια σχόλια αν θέλει. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε κατευθείαν με τις ε, παρουσιάσεις γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά οπότε θα σχολιάσω αργότερα Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε με του εισηγητές, μετά τους σκιώδεις και μετά θα ακούσουμε τα μέλη των δύο επιτροπών. Η κυρία Βίρκουνεν πρώτα, ως εισηγήτρια εκ μέρους της Ήτρα και θα μπορούσατε βεβαίως, θα μπορούσε και κάποιος, α, ο κύριος Φαμπ θα μιλήσει εκ μέρους του κυρίου Ζουβά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε ο Πρόεδρος Μπούζεκ, ο συνεισηγητή μου, ο κύριο ε, Ζουβάν, δεν είναι εδώ σήμερα δυστυχώς, αλλά έχουμε, είχαμε πολύ στενή συνεργασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ε, εβδομάδων και με τους πιο συγητές για, ε, για την έκθεση για τις online πλατφόρμες και όπως υπόθηκε ήδη έχουμε 462 τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των δύο επιτροπών που ήταν τόσο ενεργά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, όλες, σχεδόν όλες οι τροπολογίες ήταν πραγματικά πολύ θετικέ και νομίζω ότι τονίζουν τις, ε, τις ωφέλειες της, ε, των online ε, πλατφορμών, τα νέα μοντέλα, τα επιχειρησιακά, τι μπορούν να μας προσφέρουν και πόσα πολλά πλεονεκτήματα μπορεί να έχει η ευρωπαϊκή οικονομία μέσω αυτών, λόγω ακριβώς αυτών των πλατφορμών. Επίσης, οι κάποιες ε, τροπολογίες είχαν να κάνουν με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις οποίες βεβαίως συζητούμε και στις, ε, συζητήσαμε στις παλαιότερες ε, συνεδριάσεις των επιτροπών μας. Μέχρι στιγμή φαίνεται ότι το πιο δύσκολο ακαθόδε θέματα είναι το θέμα τη ευθύνη. Όπω ξέρουμε, έχουμε την σχετική οδηγία, η οποία είναι πολύ καλή και καλύπτει τα περισσότερα θέματα. Αλλά ίσω τα fake news και η ρητορική μίσους ε, τα... είναι θέματα που πρέπει ακόμα να διευκρινιστούν για το πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Ξέρω ότι όλοι είναι... Περισβεύουν ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι σημαντική ε, αξία για μας και βεβαίως δεν θέλουμε να υπάρχουν ε, περιορισμοί στην, στο ίντερνετ, αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και ανάληψη ευθύνης και για το περιεχόμενο και θα πρέπει να βρεθεί εδώ μια ισορροπία για το σημείο αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε και τις, ε... τις επόμενες ημέρες γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις αρκετά αντικρουόμενες και εντός των δύο επιτροπών μας. Οπότε, έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις ε, για 36 συμβαστικές προτάσεις και έχουμε, προετοιμάζουμε ακόμη 10. Έχουμε κάνει δύο συναντήσεις με τους Κιώδης και θα κάνουμε άλλη μία, σίγουρα και να ευχαριστήσω και όλες τις υπόλοιπες ομάδες βέβαια για το feedback που μας έδωσαν, τα σχόλια. Όλες οι ε, ομάδες δουλεύουν πολύ αποτελεσματικά γιατί πάντα χρειάζεται ε, πολλή δουλειά όταν υπάρχουν δύο επιτροπέ που συνεργάζονται για μία έκθεση. Χρειάζεται πολύ περισσότερο συντονισμό, εσωτερικό και μεταξύ των ε, ε, επιτροπών αλλά και μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Οπότε το χρονοδιάγραμμα πάντα είναι πολύ αυστηρό, όπω είναι και τώρα, αλλά ω εισηγητέ εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε με όλου του κοιόδης εισηγητέ, να ολοκληρώσουμε τι συμβαστικέ προτάσει εγκαίρω και να καταστήσουμε όσο πιο καλή γίνεται την έκθεση αυτή. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και όλα τα μέλη των Επιτροπών για τις τροπολογίες που μας έστειλαν, γιατί λόγω αυτών των τροπολογιών ακριβώς και λόγω των δικών σας σχολείων η έκθεση θα είναι πολύ καλή. Τώρα δουλεύουμε τις ε, συμβαστικές προτάσεις έτσι ώστε να έχουμε μεγάλη στήριξη. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, η ψηφοφορία θα γίνει στο Στρασβούργο στις 18 Μαΐου, που σημαίνει ότι έχουμε κάποιες εβδομάδες ακόμη ε, για να δουλέψουμε μαζί με τις ε, υπόλοιπες ομάδες και εγώ πραγματικά αναμένω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σφαμπ, εκ μέρους του κυρίου Ζουβάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έλαβα πληροφορίες καθώς και ένα σημείωμα του συναδέλφου Φιλίππε Ζουβέν που όπως ήδη είπατε δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ λόγω των χθεσινών γαλλικών εκλογών. Μου άφησε κάποια σχόλια που θα σας παρουσιάσω. Καταρχάς θέλει να συγχαρεί και να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, και όπως ε, ήδη είπε η συνάδελφος ε, του κυρία Βερκούνεν τώρα πρέπει να γίνει δουλειά για την εξέβρεση συμβιβαστικών που για την ώρα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρε ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο του τμήμα. Τα βασικά θέματα όπου διαρωτάται ο Φιλίπ είναι ακριβώς τα ζητήματα κλειδιά όπως ο ορισμός των πλατφορμών ε, και πώς θα καταφέρουμε να έχουμε έναν τέτοιον ορισμό, πώς μπορούμε να ξαναδούμε το, και κατά πόσο χρειάζεται να ξαναδούμε το καθεστώς ευθύνη των πλατφορμών που τώρα διέπεται από την οδηγία e-commerce. Τρίτον, πώς θα εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία των καταναλωτών και πώς θα εγγυηθούμε περισσότερο τη διαφάνεια και την νομική ασφάλεια για όλες τις επιγραμμικές δραστηριότητες. Τέταρτον, πώς θα ορίσουμε αυτό που η Κομισιόν ορίζει ισορροπημένο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο που ορίζει μια καλή δόση του υφιστάμενου δικαίου, αυτορύθμισης και συγκεκριμένου δικαίου για συγκεκριμένα προβλήματα και τέλος πώς θα θεσπίσουμε ένα ισότιμο πεδίο για όλους και να αποφύγουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές εναντίον των καταναλωτών και των ε, ε, επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στις 10 Μαΐου θα υποβάλει τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η ίδια ε, και άρα πρέπει να βιαστούμε ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ε, ε, παρέμβει εγκαίρως για να επηρεάσει την εργασία της Επιτροπής. Για αυτό το λόγο, ο Φιλίπ, όπως ήδη είπε η συνάδελφος Χένα, εργάζεται για να, βρούμε, να φτάσουμε σε μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου και να καταλήξουμε σε ισορροπία με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βεβαίω θα πρέπει να είναι πρακτικέ, ευέλικτε και στο πλαίσιο αυτό χρήσιμες για τις επιχειρήσεις αλλά και θα στέκουν ώστε οι ρυθμίσεις και οι νόμοι που έχουμε στην Ευρώπη να γίνονται σεβαστοί από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τους δύο. Να περάσουμε τώρα στους σκιώδεις εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και των δύο Επιτροπών να ζητήσω τον κύριο Χωσέ Μπλάνκο Λόπες να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα παρέμβω στο όνομα του συναδέλφου της ΣΥΜΚΟ, του Σέρχιο Κουτιέρεθ. Γι' αυτό και σας ζητώ να είστε λίγο διαλλακτικοί μαζί μου. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω αυτό που τονίσαμε και εγώ και ο συντροφός μου στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Οι συντάκτες έχουν ε, υποβάλει ένα καλό έγγραφο κίνηση, αλλά με μια σοβαρή έλλειψη, δηλαδή την κοινωνική διάσταση αυτής της ψηφιακής οικονομίας που δεν θίγεται καθόλου. Ε, θα, οι διάφορες δραστηριότητες στις οποίες λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες ε, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, μάλλον δεν υπάρχουν διατάξεις για τους ε, εργαζόμενους ώστε να μπορούν οι χρήστες να μπορούν να μπουν σε άμεση επαφή ε, με βάση ας πούμε για διευκρίνηση ή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται επιγραμμικά ή για κάποιο παροχή υπηρεσίες, για ανταλλαγή πληροφοριών ή για την ε, κοινοποίηση αυτών των ε, ε, ε, υπηρεσιών. Και στις διαπραγματεύσεις και τις συμβιβαστικές σε αυτό επιμένουν. Παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες για αυτή την έκθεση που εύκολα θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε τέσσερις, σε τέσσερις ομάδες οι γενικές προτεραιότητες. Πρώτον, ανάγκη νομοθεσίας. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αφού διάβασαμε λεπτομέρειες της τροπολογίας των υπολείπων ομάδων μπορούμε να συνοψίσουμε ότι συζήτηση συζήτηση που γίνεται τώρα για τις διαπραγματεύσεις των συμβιβαστικών έχουν να κάνουν με δύο βασικά θέματα. Εκείνο ε, που πιστεύουν ότι η σημερινή νομοθεσία καλύπτει πλήρως ε, τις επιγραμμικές πλατφόρμες ε, ε, και απ' την άλλη τους σοσιαλιστές και άλλους που πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες φαιές ζώνες που πρέπει να καλυφθούν. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι εδώ έχουμε ήδη κάνει εκτεταμένες συζητήσεις με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, με πανεπιστημιακούς, με εμπειρογνώμονες της Κομισιόν και ούτω καθεξής στο πλαίσιο του φόρουμ της ε, ε, συνεδρίασης εργασίας για την ψηφιακή, εργασία, ψηφιακή αγορά, με καθώς και σε σχέση με τις επιγραμματικές διαδρομικές πλατφόρμες ε, που καλύπτει αυτήν ε, την ε, τριγωνική σχέση ανάμεσα στους πλατφόρμες, τους καταναλωτές και τους παρόχους. Εδώ λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι μόνο με την αυτορύθμιση δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις υφιστάμενες νομοθεσίες που καλύπτουν τα ζητήματα του ανταγωνισμού. Ε, και που μπορεί να οδηγήσει αυτό σε ασαφείς κανόνες αλλά και σε ε, dumping, κοινωνικό dumping επιγραμμικού τύπου. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένη μορφή εξέλιξη των ισχυών των κανόνων, ώστε να υπάρξει μια ισορροπημένη και βιώσιμη εξέλιξη. Θέλουμε να ζητήσουμε από την Κομισιό να προχωρήσει σε έναν ορισμό, ώστε οι επιγραμμικές πλατφόρμες σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύονται από ταξινόμηση αυτών, που θα κάνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτού που προσφέρουν ε, και ε, πραγματική εργασία, αλλά πέρα από την εικονική, και από αυτές που ε, συμμετέχουν ε, χωρίς προσωπικό, καθώς και διάκριση ανάμεσα στις εμπορικές πλατφόρμες και τις μη εμπορικές. Σε σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα, οι ευρωπαϊκές ε, εργασιακές αγορές εξελίσσονται σε μορφές άτυπης ή μη ρυθμιζόμενης εργασίας, όπως η μη ρυθμιζομενες εργασιες οπως η αλακάρτα εργασία, η αυτόνομη ανεξάρτητη εργασία ή η ενδιάμεση εργασία για αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται για τις πλατφόρμες να έχουν ε, και κατάλληλες συνθήκες εργασίας, γιατί γίνεται εκτεταμένα περισσότερη χρήση του αυτόνομου και ανεξάρτητου εργαζόμενου από πλευρά αυτών των πλατφορμών. Γι' αυτό η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίσει σε ποιο βαθμό η ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να ισχύσει και για την ψηφιακή αγορά εργασίας και πόσο θα εγγυάται την ε, προσαρμογή και την τήρηση αυτή τη νομοθεσία. Πιστεύουμε οι σοσιαλιστές ότι η παιδεία και η το καινοτομία είναι απαραίτητε για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με επιτυχία να ανταγωνιστεί στι παγκόσμιε αγορέ, διατηρώντα ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόληση και συνθήκε ισότιμε. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι υδροποδολογίες ώστε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλες τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις μάλλον που προσφέρουν υπηρεσίες ανεξάρτητα αν αυτές προσφέρονται επιγραμμικά ή όχι. Και να εγγυάται ότι όλες οι εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών θα πληρώνουν τις φόρους τους στο μέρος όπου δημιουργείται το οικονομικό κέρδος λόγω της δραστηριότητάς τους. Και για τους σοσιαλιστές είναι προφανές ότι υπάρχουν πλατφόρμες που παίζουν ρόλο πιο δραστήριο από ότι απλώς ενδιάμεση. Γι' αυτό η σημερινή νομοθεσία θεωρούμε ότι δεν αρκεί και γι' αυτό έχουμε παρουσιάσει και μεταξύ άλλων μια πρόταση ώστε να ζητήσουμε γρήγορη διαδικασία για την ε, εντοπισμό των, του περιεχομένου που δεν σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα ε, σε άλλες δεν τρο... Ο πρόεδρος διακόπτει. Α, ένα λεπτό ακόμα παρακαλώ πρόεδρε, γιατί μιλώ και στο όνομα του συναδέλφου. Ναι, αλλά έχετε μιλήσει έξι λεπτά σχεδόν. Ναι, ναι, μόνο ένα λεπτάκι ακόμα σας ζητώ. Στις, ε, στη 224 και 225, 26, 27. Ζητάμε να τεθεί στη διάθεση των χρηστών ε, εργαλείο ώστε να μπορούν να διακρίνουν τις ψευδείς ειδήσει που κυκλοφορούν σε αυτές τις πλατφόρμες καθώς και την απαγόρευση ε, λόγου μίσους. Ε, τώρα έχουμε τον κύριο Ντάνιελ Ντάλτον από την ΙΜΚΟ. Oh. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρους και των δύο ε, και της συναδέλφου. Όπως ε, έχουμε ξαναπεί και εγώ και η Άνελίν, από τη δική μας την ε, πλευρά πρέπει να επικεντρωθούμε στο θετικό περιεχόμενο για, την, ε, για τον κλάδο αυτό, για την οικονομία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπλεκούμε με τις διάφορες, τις διάφορες τομείς της νομοθεσίας. Πρέπει να δούμε πού εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες, αλλά δεν είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι οι online πλατφόρμες δεν ταιριάζουν στους υπάρχοντες κανόνες επειδή είναι επιχειρησιακά μοντέλα. Ε, νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Δεν συμφωνούμε με αυτή την ε, υπόθεση. Επίση, δεν συμφωνούμε ότι υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν καταλαβαίνω ακριβώ τη θέση αυτή, γιατί πολλέ πλατφόρμε έχουν επιτύχει παρά το γεγονό ότι υπάρχουν ακριβώ αυτοί οι κανόνε που έχουν ε, δημιουργηθεί για να προστατεύουν του ανταγωνιστέ του. Οπότε δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Το ίντερνετ έχει ε, επιφέρει περισσότερη δημοκρατία στον κόσμο και δίνει περισσότερα δικαιώματα στους ε, ε, καταναλωτές και στους εργαζόμενους όσο δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στην ιστορία. Είναι πολύ καλό λοιπόν αυτό. Είναι καλό για τις εργασιακές συνθήκες γιατί έτσι αφαιρείται η ισχύ από τους εργοδότες και πηγαίνει στους εργαζομένους. Δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν να πηγαίνουν στη γραφείο από τις 9 μέχρι τις 5 μέχρι τα επόμενα, για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια. Μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο τη ζωής τους. Και αυτό είναι καλό. Επιτρέπει στους πολίτες να έχουν να έχουν δυνατότητα ε, δραστηριότητας επαγγελματικής ε, και που δεν υπήρχε παλιά τέτοια δυνατότητα. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ ε, δυνατότητε για άτομα που δεν είχαν καμία εξουσία παλιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πού είναι ακριβώ το πρόβλημα. Τώρα, για κάποια συγκεκριμένα ε, στοιχεία, για τον ορισμό των πλατφορμών, δεν βλέπω την ανάγκη ή τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ακριβή ορισμό συνολικό. Η πλατφόρμα θα πρέπει να ρυθμίζεται όπω γίνεται, ανατομέα, όπω γίνεται και τώρα δηλαδή και δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται και δεν είναι και σημαντικό νομίζω να υπάρξει ορισμός των, των πλατφορμών. Επίσης συμφωνώ με την διευκόλυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει κάνοντας την Ευρώπη ένα καλό περιβάλλον ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι πλατφόρμες, όλα αυτά τα προστατευτικά μέτρα που υπάρχουν, απλώς ε, ωφελούν τους υπάρχοντες παρόχους. Οπότε ε, να μην υπάρχει ανταγωνισμός, να υπάρχει καινοτομία, ε, δημιουργία, να προστατεύσουμε τις ε, πλατφόρμες στην Ευρώπη και να ενισχύσουμε τους καταναλωτές. Για την ευθύνη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι πλατφόρμες βεβαίως πρέπει να, την, να τηρούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με τους ασφαλείς λιμένες των ενδιαμέσων που είναι απαραίτητη για, την, για τον ανοιχτό χαρακτήρα του ίντερνετ, για την νομική βεβαιότητα και την αποφυγή παρεμβάσεων. Επίση, υπάρχει και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι κανόνες που υπάρχουν εκεί πρέπει να ε, εξεταστούν και για το μέλλον πρέπει να υπάρχει, στην έκθεση υπάρχουν πολλές θετικές ε, ε, ε, απόψεις για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εξελίξουμε την εμπιστοσύνη, αλλά όταν μια πλατφόρμα χάσει την εμπιστοσύνη, χάνει και τους πελάτες της. Αυτό είναι το καλό με την ψηφιακή οικονομία. Και επίσης με την συνεργατική οικονομία κάνει τον καταναλωτή βασιλιά, όπως δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα για τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την έκθεση, για την φορητότητα για, την, ε, για τις ροές δεδομένων διασυνοριακά που είναι πολύ σημαντικές για τις ε, ε, ε επιχειρήσεις που λειτουργούν διασυνοριακά έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλέ σχέσει και με του εμπορικού μα εταίρου σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρώπη ω ε, ε, ε, λιμένα πληροφοριών να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Είναι πολύ χρήσιμη η βάση λοιπόν που έχουμε για να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ πολύ του συζητητέ που μα έφτασαν σε αυτή, την, σε αυτή τη φάση που ούτω ή άλλω ήταν δύσκολο να φτάσουμε και χαίρομαι που θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδο στην έκθεση αυτή τι επόμενε εβδομάδε. Ξέρω ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμη, αλλά θα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μέσα τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Από την Άλντε. Από την Άλντε λοιπόν και από τις δύο ε, επιτροπές η κυρία Κάλας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έξι λεπτά γιατί θα μιλήσω εξ ονόματος και των δύο σκιώδων, επειδή ξέρω ότι είσαστε και αυστηρός με τον χρόνο. Πρώτα λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές για την εργασία τους, για τη σύνταξη εκθέσεως καθώς και για τις τροπολογίες που έχουμε ήδη λάβει και τις οποίες επεξεργαζόμαστε. Πολλά θετικά στοιχεία βρίσκω στις συμβαστικές τροπολογίες που αναγνωρίζουν τον ρόλο των πλατφορμών που δημιουργούν ευκαιρίες και για τους καταναλωτές, υπέρ των καταναλωτών δηλαδή και υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εξετάζουμε και διάφορα θέματα σε σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την διαφάνεια ε, συστημάτων franchising και άλλα σχετικά. και για ε, άλλες επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στις πλατφόρμες για να αναπτυχθούν. Κάποιες διαφορές έχουμε βέβαια ακόμα σε ορισμένες συμβαστικές τροπολογίες και πρώτα η Άλντε προτιμά να εξετάσει τα ζητήματα εφαρμογής πριν να ζητήσει και άλλη νομοθεσία. Πολλά νομοθετήματα επικαιροποιούνται για την ώρα και θα προτιμούσαμε η έκθεση να ζητήσει νέα νομοθεσία μόνο εφόσον ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Και ε, για τις πλατφόρμες νομίζουμε ότι η νομοθεσία ε, δεν, δεν θα έπρεπε να ορίζει ποιε είναι αυτές. Και η, γενική, αρμόδια γενική διεύθυνση θα πρέπει να εξετάσει πώς θα αντιμετωπίσει τις νέες μορφές επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν τις αγορές ε, μέσα σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν τις επιπτώσεις των δεδομένων και θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες για να λαμβάνουν αποφάσεις. Ε, δεν συμφωνούμε όμως απολύτως με τα όσα λέει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Και τέλος, το ζήτημα της ευθύνης των επιγραμμικών πλατφορμών. Υπάρχουν και ορισμένε παράγραφοι, οι οποίε αναφέρονται όλες στο ίδιο θέμα, αλλά με διαφορετικές διατυπώσεις και έτσι προκαλείται σύγχυση. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τις πλατφόρμες, για τις παραγράφους που εξετάζουν την ευθύνη των πλατφορμών μόνο από την πλευρά των επιχειρήσεων που διαθέτουν copyright και όχι μόνο από την άψη των χρηστών, αλλά ιδίω για θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών. Και δεν είναι και κανένα μικρό πράγμα αυτό, διότι μιλούμε για ελευθερία εκφράσεως, για προστασία δεδομένων και πληροφοριών και πιο συγκεκριμένα για τις παραγράφους αυτές. Τι είδους περιεχόμενο θέλουμε να είναι υπεύθυνε, ε, ε, γι' αυτό δηλαδή, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αρχίσουν να εξετάζουν πιο περιεχόμενο επιβλαβές και ούτω καθεξής. Ε, τότε καλύτερα να πούν σε επιχειρήσεις να μην αρχίσουν καν να δραστηριοποιούνται. Ως πολιτικοί γνωρίζουμε βεβαίως ότι γίνονται και πάρα πολλά σχόλια σε βάρος μας στις πλατφόρμες. Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα κρίνει τι είναι ενδεδειγμένο και τι όχι. Η πολιτική μου ομάδα ε, δέχεται μονάχα την αναφορά σε παράνομες παράνομο περιεχόμενο, εφόσον δηλαδή οι πλατφόρμες ε, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει παράνομο περιεχόμενο και δεν το αφαιρούν. Δεύτερο, για τα προληπτικά μέτρα. Ζητούμε από τις πλατφόρμες να προλαμβάνουν περιεχόμενο με χαρακτήρα μη κατάλληλο κλπ. Υπάρχουν εθελοντικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι πλατφόρμες για παράνομο περιεχόμενο, δηλαδή να έχουν σαφέστερες ε, διατάξεις για το ε, πιο περιεχόμενο επιτρέπεται ή όχι, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει μια γενική υποχρέωση εποπτείας και εφαρμογή φίλτρων. Επίσης, για την, για την παράνομη χρήση δεδομένων ατόμων. Οι αλγόριθμοι δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι σωστό και τι όχι, τι μπορεί να σημαίνει ηρωνία, τι μπορεί να σημαίνει παραβία και ούτω καθεξής. Όπως είπα και στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Επειδή οι περισσότερες πλατφόρμες δεν είναι καν ευρωπαϊκές, αλλά αμερικανικές ή ρωσικές ή κινέζικες, διερωτώ με γιατί οι εισηγητέ με τόση άνεση ζητούν από μη ευρωπαϊκές εταιρείε να ε, φιλτράρουν περιεχόμενο που παράγουν Ευρωπαίοι παραγωγοί χωρίς ε, να σκέφτονται τις επιπτώσεις. Ε, να εξετάζουν λοιπόν και τα συστήματα που λέγονται notice και down και ταυτόχρονα και ρίτες προφύλαξης για τους χρήστες, αλλά δεν θα δεχτούμε διατυπώσεις οι οποίες να υπονομεύουν ολόκληρο το πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ευχαριστώ. Μισελ Ραϊμό. Των πρασίνουν. Θα μιλήσει ο συνάδελφό μου εκ μέρου μα. Ή συνάδελφό μα, κυρία Ρέντα. Σα uh, Σας ευχαριστώ. Όπως είπε ο συνάδελφός μου, θα μιλήσω εξ ονόματος και των δύο επιτροπών, αφού πρώτα ευχαριστήσω τους εισηγητές για το δεύτερο αυτό πακέτο συμβαστικών τροπολογιών που ε, περιέχει σημεία που μπορούμε πιο πολύ να συμφωνήσουμε αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά εκκρεμή θέματα. Πρώτα, θέλουμε να τονίσουμε και πάλι ότι για την παρούσα έκθεση βλέπουμε τη θεμενεξία είναι σημαντικό να στοχεύσουμε σε τομεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη προωθήσει νομοθεσία. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχουν παράγραφοι, για την οδηγία EBMS που η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πρόκειται να ψηφίσει την έκθεση και ιδίω για θέματα ευθύνη. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε και πάλι ότι η οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να αποτελεί την βάση για όλε τι διαβουλεύσει μα και χαίρομαι που ο εισηγητής μίλησε για την σημασία της ε, οδηγίας ηλεκτρονικού εμπορίου για το περιβάλλον του διαδικτύου. Ιδίω δεν υποστηρίζουμε οποιαδήποτε αναφορά στην ενίσχυση της εποπτείας monitoring, διότι θεωρούμε ότι αυτό αντιβαίνει και στο περιεχόμενο της ε, οδηγίας ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που έχει τονίσει ότι τέτοια γενική εποπτεία, γενική παρακολούθηση παραβιάζει και την ελευθερία έκφρασης των προσώπων και των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά ορισμένε από τι νέε προκλήσει σχετικά με hate speech και fake news, ήδη έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ για τα πράγματα αυτά και στι χώρε μέλη, οι οποίε έχουν κάνει κάποιε απόπειρε να προωθήσουν κάποια νομοθετική ρύθμιση. Αλλά το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, στις, ε, που έχουμε εντοπίσει μάλλον στι ε, συζητήσει αυτέ, είναι ότι τα περισσότερα από τα μηνύματα μίσους κλπ. δεν είναι στην πραγματικότητα παράνομα υπό την ισχύ του δικαίου των χωρών μελών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με αριθμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης, μόνο 15% όλων των μηνυμάτων μίσους είναι πραγματικά παράνομα σύμφωνα με τα εθνικά δίκαια. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι η ευθύνη μπορεί να είναι το σωστό εργαλείο, διότι αν το περιεχόμενο ούτω ή άλλω δεν είναι παράνομο, είναι πολύ δύσκολο να ζητήσετε από μια πλατφόρμα να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για το περιεχόμενο αυτό. Ίσως είναι πιο χρήσιμο να αντιμετωπιστεί η καταλληλότητα των νομικών ποινικών προβλέψεων στις χώρες μέλη. Υπάρχει και το θεμελιώδες πρόβλημα ότι διαφορετικοί τύποι περιεχομένου αλλά και, παρά, και παράνομο ενδεχομένω περιεχομένου μπορεί να χρειάζονται διαφορετικέ αντιμετωπίσει και επομένω θα χρειαστούν νομοθετικέ ρυθμίσει. Και το notice and take down regime μπορεί να είναι και το πιο κατάλληλο μέσο γιατί θα δώσει περισσότερη σαφήνεια στις πλατφόρμες σχετικά με το ποιε υποχρεώσεις υπάρχουν για ποια είδη περιεχομένου. Για παράδειγμα, για μηνύματα μίσους και fake news ψευδή νέα είναι μη επιθυμητό περιεχόμενο είναι κάτι άλλο. Για το ζήτημα των παραβιάσεων copyright δεν είναι ακριβώς το περιεχόμενο που είναι παρανομό, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται, εφόσον για παράδειγμα δεν υπάρχει εξαίρεση από το copyright. Και εκεί αυτόματα μέτρα δεν μπορούν να το καθορίσουν αυτό. Υπάρχουν και άλλα πλαίσια, για παράδειγμα, η αφαίρεση εικόνων κατάχρησης ε, ή κακοποίησης παιδιών που δεν θέλετε να ειδοποιήσετε το υποκείμενο που τα έχει αναρτήσει τα πράγματα αυτά ότι ε, παρακολουθείτε διότι δεν θέλετε να παρέμβετε στο έργο των διοκτικών αρχών. Μια πρόταση λοιπόν η οποία θα θεσπίζει διαδικασίες για notice and take down θα πρέπει να περιλαμβάνει και counter notice διαδικασίες και ποιες είναι οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν τότε οι πλατφόρμες. Ε, αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο να προβλεφθεί. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που βλέπουμε με το σχέδιο συμβαστικών τροπολογιών. Αναφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιοκτησία των δεδομένων. Έχει μείνει ανοιχτό το ερώτημα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνδεσιμότητα, όπου είχε προτείνει έξι διαφορετικές επιλογές πολιτικής και μόνο μία από αυτές περιλάμβανε το δικαίωμα κυριότητας που νομίζουμε ότι είναι λάθος προσέγγιση. Είναι καλύτερα να υπάρξει μια ειδική συμβαστική τροπολογία που να αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτή και να περιλαμβάνει τη σύσταση του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, θέλουμε να υποστηρίξουμε default contact, contract rules, κανόνες δηλαδή ε, για σύμβαση σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τίποτε, για τα διάφορα σημεία διατομής κλπ. Και να το δούμε σε αυτό το πλαίσιο, όχι να το πούμε χωρίς πρώτα να έχει συζητηθεί εάν συμφωνούμε ή όχι με την ιδέα αυτή. Τέλος, οι συμβαστικές τροπολογίες για ζητήματα διαφάνειας και εντιμότητα σε, διαδικασία, σε, ε, σε, σε σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Συμφωνούμε με την γραμμή που ακολουθούν οι συγητές, αλλά συνολικά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που χρειάζεται να γίνει στις συμβαστικές τροπολογίες, ώστε να ικανοποιούμεθα. Ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Εδώ λίγη ο κατάλογος των σκιωδών. Και θα, θα παραχωρήσω τα ενία της συζητήσεως στην κυρία Πίκη Φόρντ. Ορισμένοι έχουν ζητήσει το λόγο. Νίκολα Ντάντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς Καταρχάς, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι το θέμα της ε, ευθύνης ε, ε, τονίστηκε πολύ καλά από την εισηγήτρια. αυτή είναι η πραγματική πρόκληση. Είμαστε ενώπιον ενός κόσμου που δεν γνωρίζουμε εις βάθος και που είναι περίπλοκος να τον κατανοήσει κανείς, αλλά που διαπερνά την καθημερινότητά μας, διεισδύει στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ίσως τις, υποχρεώσει τη παραδοσιακή ε, οικονομία από αυτέ τη ψηφιακή. Ε, θα έχουμε ευθύνε και υποχρεώσει και στην ε, ψηφιακή οικονομία και πρέπει να ελέγξουμε και την αξιοπιστία των πλατφορμών αυτών. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερου κανόνε, αλλά καλού κανόνε Και το γεγονό ότι διαρκώ παραπέμπουμε στην οδηγία e-commerce είναι σωστό, αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί αυτή ασχολείται με την ανταλλαγή των προϊόντων και όχι των υπηρεσιών. Μιλάει για ένα σωρό πτυχέ, αλλά όχι για όλε τι πτυχέ με τι οποίε ασχολούνται σήμερα οι πλατφόρμες που περιλαμβάνουν ένα σωρό πτυχέ τη ζωή μας. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε οι πλατφόρμες να έχουν διαφορετικέ και ε, διακριτικέ στάσει απέναντι στους ε, χρήστε και του κατανολωτέ. Είναι κάτι που υπάρχει ήδη. Δείτε στη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τη συζήτηση, όπου η εξέλιξη των πλατφορμών έχει προχωρήσει περισσότερο και τώρα συζητάτε πόσο και αν μπορούν οι πλατφόρμε να παίξουν ρόλο διακρίσεων για ορισμένες κοινωνικές τάξεις. Πιστεύω πως πρέπει σε αυτό το θέμα να δουλέψουμε και για την ευθύνη το, την ε, εκδοτικού τύπου ε, των πλατφορμών σε σχέση με τις ειδήσει που παρουσιάζουν και προβάλλουν και εδώ. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική και με την ελευθερία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλές από τις δραστηριότητες και τις πολιτικές γνώσεις των ανθρώπων περνούν τώρα από τις πλατφόρμες και αυτό επηρεάζει άμεσα τα δημοκρατικά συστήματα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ενώπιον αυτών των προκλήσεων οφείλουμε να έχουμε μια στάση υψηλής ευθύνη και να προσπαθήσουμε να αδράξουμε τις ευκαιρίες βεβαίως που προσφέρουν οι πλατφόρμες, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να εντοπίζουμε τις ευθύνες που επιβαρύνουν τον καθένα και είναι ουσιαστικό στοιχείο της κάθε οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ. Υπάρχει πολύ δυναμικό στις online πλατφόρμες γιατί προσφέρουν νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Δίνει στους, ε, στους καταναλωτές μια επιλογή και ενισχύουν τον ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, το μερίδιο της, ε, στην Ευρώπη ε, των επιγραμμικών πλατφορμών είναι πολύ μικρό και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε αν θέλουμε όντω να φτάσουμε τους εταίρους μας στη ΣΥΠΑ και στην Ασία. Υποστηρίζω τι τροπολογίε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δυναμικό της αύξησης των ε, επιγραμμικών πλατφορμών στην Ευρώπη και κυρίως την ε, ε, ανάγκη για εξειδικευμένους εργαζόμενους για τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Επίσης για, την, για τις για την ευθύνη των ενδιαμέσων στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίση, η τεχνολογικώ ουδέτερη προσέγγιση που είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να μην αποτρέψουμε οποιασδήποτε μελλοντικέ προσπάθειε να πραγματοποιηθούν. Επίση, υποστηρίζω τι ε, τροπολογίε των συναδέλφων που λένε ότι οι πλατφόρμε ορίζονται καλύτερα ανατομέα, σε τομιακή ε, νομοθεσία ανάλογα με τις ε, υπηρεσίες που προσφέρουν, αντί να δημιουργήσουμε ένα συνολικό γενικό ορισμό. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε παλαιότερες μεικτές συνεδριάσεις, υπάρχουν ε, πλατφόρμες που παρέχουν ε, ε, υποδομές, ενώ άλλες παρέχουν υπηρεσίες. Οπότε δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία λύση για όλες τις πλατφόρμες, γιατί αν γίνει αυτό θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κοινοτομία και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να μην επηρεάσουμε αρνητικά την κοινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης καλωσορίζω τις ε, τροπολογίες που τονίζουν την ευθύνη των ε, πλατφορμών να δημιουργήσουν αυτορυθμιστικά μέτρα ώστε να αποτρέψουν το παράνομο περιεχόμενο και τα αγαθά. Παρόλα αυτά χωρίς να, ε, να υποβιβάζουν τα δικαιώματα της έκφρασης και γενικώ τα δικαιώματα των καταναλωτών. Πολλές επιγραμμικές πλατφόρμες ε, ε, ασχολούνται με το θέμα της ε, ε, αναθεώρησής τους, αναδόμησής τους. Θεωρώ ότι πολύ καλό θα ήταν να δούμε τι γίνεται με τους κανόνες για τον, για τον θέμα του ανταγωνισμού που υπάρχουν από τις οδηγίες. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια νέα αρχή ευρωπαϊκή για να αξιολογήσουμε και να ελέγξουμε τα συστήματα αυτά αναθεώρησης των επιγραμμικών πλατφορμών όπως προτείνουν κάποιες, κάποιες τροπολογίες. Συνολικά είναι καλή η έκθεση και ε, μπορώ να υποστηρίξω πολλές από τις τροπολογίες. Καλή επιτυχία στους ε, εισηγητές και στους χειώδες που, και τη μελλοντική δουλειά τους που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές για την εργασία τους. Όλη η οικονομία των ε, πλατφορμών βασίζεται στην ε, αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές της ε, λόγω πλατφόρμας. Όταν κανείς ρωτήσει τους Ευρωπαίους σήμερα, μόνο 22% έχουν εμπιστοσύνη στις πλατφόρμες και γενικότερα ευρύτερα στα δίκτυα εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι να ενισχύσουμε αυτή την πίστη στις πλατφόρμες και την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, πράγμα που περνά από διάφορα στοιχεία, εκ των οποίων ορισμένα αναφέρθηκαν, ε, ευθύνη, δέσμευση, των πλατφορμών, κάποιες φορές με κάποιες υποχρεώσεις για εκείνες, δηλαδή υποχρέωση να δίνουν πληροφορίες στους καταναλωτές, ε, ε, ε, να δίνουν πληροφορίες για το δίκαιο, το δίκαιο της εργασίας, στο εργατικό δίκαιο. Ε, περνά επίσης από πιο στενή συνεργασία μεταξύ πλατφορμών και διοίκησης ε, του εκάστοτου κράτους, αλλά επίσης θέλω να επιστήσω την προσοχή στα σχόλια που γίνονται ε, στις πλατφόρμες ε, όσον αφορά την φήμη αυτών των πλατφορμών. Θα ήθελα πραγματικά εδώ να στρατευθώ για τη δημιουργία ε, μηχανισμών πιστοποίησης αυτών των σχολείων, να ξέρουμε δηλαδή από πού προέρχονται πραγματικά θα πρέπει να βρεθεί μια ανισορροπία, γιατί αυτό που έχει σημασία και πρέπει να το θυμίσουμε είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσει κανείς την δυναμική ανάπτυξη και καινοτομία των πλατφορμών αυτών. Ευχαριστώ. Εντουάρτ Μάρτιν. Μαχτά. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγο ο κύριο Μπούζεκ αναφέρθηκε στι γαλλικέ εκλογέ που έγιναν χθε, στον πρώτο γύρο δηλαδή των γαλλικών εκλογών και όλοι θα γνωρίζετε τα αποτελέσματα και αυτό θα πρέπει να μα κάνει να διερωτηθούμε κυρίω όταν εργαζόμαστε για τέτοια θέματα. Η ιδέα που εγώ υπερασπίζω είναι ότι πρέπει πάντοτε να μετρούμε τις αρνητικές επιπτώσεις γιατί η Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Αγορά ε, ε, με βρίσκει σύμφωνο, Όμω, πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για το πλεονέκτημα για τον πελάτη. Θα ήθελα όμω να μα προβληματίσει είναι, ποια είναι τα ωφέλη για τον πολίτη, ποια θα μπορούσαν να είναι τα ωφέλη για τον εργαζόμενο, γιατί αυτό οδηγεί στο να αγαπά κανεί ή να απεχθάνεται την Ευρώπη. Γιατί αν πίσω από αυτή την ιδέα είναι να υπάρχει ακόμα πιο έντονο ανταγωνισμό, ξέρουμε αυτό που οδηγεί αυτό ξέρουμε που μας οδηγεί η οργή των Ευρωπαίων πολιτών. Ναι, στην νέα αγορά, αλλά προσπαθεί, προσοχή το πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποια εργαλεία θα έχουμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε για κοινωνική εναρμόνιση, για φορολογική εναρμόνιση, γιατί πολλοί συνάδελφοι είπαν και κριτικάρουν συχνά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που κάνουν, λέει, κοινωνικό τουρισμό. Ναι, αλλά οι επιχειρήσεις που κάνουν φορολογικό τουρισμό, επίσης δεν έλαβε πολλά λόγια και προσοχή, το είδαμε στο παρελθόν. Μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείε ε, τηλεπικοινωνιών, όλες χωρίς εξαίρεση, μετακίνησαν ε, τις πλατφόρμες ε, κλήσεων στην Ασία ή στην Αφρική. Η καλύτερη απόδεση είναι αυτή που τους ενδιαφέρει και κυριαρχεί επί όλων των άλλων και πολλοί επενδυτές σίγουρα θα πάνε να βρουν στην πλανήτη τα σημεία που είναι τα φθηνότερα των φθηνότερων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ας κάνω κάποια σχόλια, μια που δεν μίλησα πριν. Να ευχαριστήσω τους συζητητές για την δουλειά που κάνουν για τις συμβαστικές προτάσεις. Είναι καλό να βλέπουμε τη γενική εικόνα και να θυμόμαστε ότι υπάρχει η νομοθεσία που ε, μπορεί να καλύψει πολλά από όσα συμβαίνουν στην κοινότητα των πλατφορμών συνολικά. Οπότε είναι σημαντικό η νομοθεσία που θα ζητήσουμε να εκπονηθεί να μπορεί να συνδυαστεί με τους υπάρχοντες κανόνες. Για παράδειγμα, εφαρμόζουμε την οδηγία για την προσοχή των δεδομένων, την εφαρμόζουν οι, εφαρμόζουν οι ε, εταιρείε νέε οδηγίε για την ε, ασφάλεια των πληροφοριών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην ε, θολώσουμε τα νερά. Πρέπει τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Και Κάποιες από τις συμβαστικές προτάσεις, ε, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουν απόλυτη ε, σαφήνεια σε αυτό. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς προς τους οικονομικούς ε, εμπλεκόμενους φορείς, ότι υπάρχει η νομοθεσία και ότι αυτή που θα εγκριθεί ή μόλις εγκρίθηκε μπορεί να συνδυαστεί με την παλιά. Τώρα για το θέμα της ευθύνης των ενδιαμέσων. Αυτό καθορίζεται από την οδηγία για, την, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και είναι σαφή η οδηγία και είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς ε, operators γιατί ξέρουν ποιε είναι οι ευθύνε τους. Έγιναν επίσης κάποια ξεκάθαρα σχόλια για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι operators, ε, οι πάροχοι, αν τους συζητήσουμε να αντιδράσουν σε πράγματα που ούτως ή άλλως δεν είναι ορισμένα ως ε, παράνομα. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, στο τι αλλαγέ θα κάνουμε στην ευθύνη των ενδιαμέσων, γιατί μπορεί όντως να αποσταθεροποιήσουν άλλα κομμάτια της ψηφιακής αγοράς και να καθυστερήσουν την καινοτομία. Είναι πολύ καλή λοιπόν η δουλειά που κάνετε για να καταλήξουμε στις συμβαστικές προτάσεις. Θα δούμε και τα όσα είπαμε στην, για την έκθεση Κάλλας Γκέπχαρτ που είχε πραγματικά έτυχε τεράστια στήριξη από τις από τις δύο επιτροπές μας και έδωσε ένα σαφές μήνυμα πριν από ένα περίπου χρόνο. Και επίση όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι, το είπε ο Νίκολα Ντάντη στην έκθεση του για την συνεργατική οικονομία. Πρέπει λοιπόν όσα έχουν υποθεί να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αντίκεινται το ένα στο άλλο. Αυτά λοιπόν είναι τα δικά μου σχόλια. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο από την Κομισιόν να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θυμίσω λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ή κινείται η πολιτική είναι, για τις πλατφόρμες είναι η πολιτική για την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία θέλουμε να ανθίσει και να μπορέσουμε να έχουμε τα ωφέλη της, σε ό,τι αφορά ε, την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, την κοινοτομία κτλ. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Επίσης ε, θέλουμε να έχουμε νέες ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Μία από του, ένας από τους βουλευτές μίλησε για το χαμηλό ποσοστό των ευρωπαϊκών ε, ε, πλατφορμών και δεν πρέπει να δημιουργήσουμε νομικά πλαίσια τα οποία καθιστούν αδύνατο για νέες, να δημιουργηθούν νέες ε, πλατφόρμες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστή ανάλογη προσέγγιση, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες πλατφόρμες. Θέλουμε, θέλουμε να έχουμε μια καλώ λειτουργούσα πλατφόρμα και για την οικονομία, για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και, την οποία να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι καταναλωτέ και οι χρήστε και οι επιχειρήσεις, γιατί όντως υπάρχουν πολλά ωφέλη. Όσο και να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από το ότι όντως οι πλατφόρμες αποτελούν ε, τον ε, ε, θεματοφύλακα των πληροφοριών των εταιριών. Το βασικό λοιπόν για μας είναι η εμπιστοσύνη. Αναφέρθηκε ήδη από εσάς το θέμα αυτό. Η εμπιστοσύνη πάντα σχετίζεται με τη διαφάνεια, σχετίζεται με τη δικαιοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και των πλατφορμών, τη σχέση δηλαδή αυτών των δύο και που τη μελετούμε τώρα και βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να εξασφαλίσουμε ότι η ελευθερία για την εξαγωγή επιχειρησιακών δραστηριοτήτων θα πρέπει να υπάρχει και για τις επιχειρήσεις και για τους χρήστες και για τις μικρές επιχειρήσεις και πλατφόρμες για να μην ε, εμποδίσουμε την καινοτομία, για να λύσουμε πραγματικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευθύνη, πολύ σημαντικό θέμα, όπως υπόθηκε και από εσάς, μιλούμε για παράνομο περιεχόμενο, όπου η νομοθεσία μπορεί να παρέμβει. Και είναι και το επίκεντρο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η στιγμή που θα περάσουμε στο επιβλαβές αλλά όχι, ε, παράνομο ε, περιεχόμενο, εκεί θα μπούμε σε πολύ αχαρτογράφητα νερά. Και τέλος, ο ορισμός, το θέμα του ορισμού των πλατφορμών. Είμαστε αρκετά συντηρητικοί ως προς αυτό, αρκετά σκεπτικοί ε, για να υπάρξει ένας ενιαίος ε, ε, ορισμός μπορεί να είναι αντιπαραγωγικός και πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Οπότε συνολικά και εν κατακλείδη πρέπει να έχουμε μια ευέλικτη, ανάλογη ανταπόκριση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αλλά ας μην πάμε πολύ μακριά. Ευχαριστώ. Θέλουν οι συγκητές να κάνουν κάποια καταληκτικά σχόλια. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε το επόμενο, το επόμενο το μισό της ε, συνεδριασής μας, οπότε έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, οπότε να ευχαριστήσω και εγώ όλους για τα σχόλιά σας. Πολύ καλές οι παρεμβάσεις σας και βλέπω ότι κανείς ε, δεν είναι δυστυχής, ακόμα τουλάχιστον με τις ε, συμβαστικές μας προτάσεις, οπότε ξέρω ότι έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε, αλλά όλοι θέλουμε να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό, ε, στην Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό είναι ο βασικό μα στόχο. Βεβαίω υπάρχουν διάφορε απόψει για το ποια είναι τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τον επιτύχουμε, πώ μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό και διαφάνεια για τι ε, πλατφόρμε. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην υπερρυθμίσουμε την Ευρώπη γιατί όλοι ε, συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε την καινοτομία στην Ευρώπη. Και εγώ είμαι αρκετά σκεπτική ό,τι αφορά την αυτορύθμιση γιατί πιστεύω ότι και τα παραδοσιακά μέσα κάνουν πολλά σε ό,τι αφορά την αυτορύθμιση, αλλά η, δεν νομίζω ότι είναι προς όφελος των πλατφορμών να δημιουργηθεί έλλειψη εμπιστοσύνη. Πρέπει να μπορούν να τι εμπιστευτούν οι καταναλωτέ. Υπάρχουν ε, κανόνε και υπάρχει νομοθεσία έτσι, και πρέπει να δούμε απλώ πώ θα την εφαρμόσουμε πριν προτείνουμε οτιδήποτε καινούριο σε επίπεδο νομοθεσία. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου για τα σχόλιά σα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα πραγματικά και, θα... και περιμένω να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά έτσι ώστε στο τέλο να μπορέσουμε να του έχουμε όλου ευχαριστημένου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, οι τροπολογίες, οι συμβαστικές προτάσεις θα μελετηθούν στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής 18 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ όλους, ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Η ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ΙΜΚΟ πάει στο 3G3. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ και θα αρχίσουμε σε λίγο. Για μας είναι πιο εύκολο εδώ στην Ήτρα.